ζητήματα που εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και στους φορείς στους οποίους απευθύνονται. Η συνεδρίαση λίγη. Καλή υπόλοιπη εβδομάδα αγαπητοί συνάδελφοι.